ενθαρρύνουν κυβερνήσεις που παραβιάζουν τους κλιματικούς κανόνες και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. η πρωτοβουλία της κομισιόν για νομοθετική πρόταση το 2021 στην πραγματικότητα βάζει προϋποθέσεις ώστε να μην φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικά κριτήρια και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίτροπε. όμως ξέρετε ο αμαζόνιος είναι δίπλα είναι εδώ. ο πλανήτης είναι μια γειτονιά όπως δυστυχώς απέδειξε και η πανδημία του covid. 19 για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε την πίεση στην κυβέρνηση της βραζιλίας και στις αρχές της περιοχής ώστε να λάβει όλα τα μέτρα για αυτό το σπουδαίο πνεύμα του κόσμου για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο Νάτσο Η έλλειψη δημοκρατίας ε, οδηγεί πάντα σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ε, πάντα οι αυταρχικές τάσεις έχουν και αυτό το πρόσωπο ε, και κινδυνεύουν οι φυσικοί πόροι από τους δημαγωγούς λαϊκιστές πολιτικούς όπως ο Μπολσονάρο, Τραμπ και άλλοι. Ουσιαστικά θέλουν τα πάντα να υπο ταχθούν ε, στη λογική της οικονομίας, στη λογική του κέρδους. Σαν το περιβάλλον ή οι συνέπειες των περιβαλλοντικών πρακτικών να μπορούσαν να περιορίζονται στα εθνικά σύνορα και βλέπουμε αυτό τον περιβαλλοντικό εθνικισμό ε, σε όλο το, το μεγαλείο σε αυτές τις χώρες και είδαμε και τα αποτελέσματά του και στην Αρκτική τα βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά και αλλού. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για πόρους, φυσικούς πόρους που αποτελούν ε, το, φυσικό τόπο διαβίωσης αυτοχθόνων ε, πληθυσμών, τους οποίους τους εκδιώχνουν από τη χώρα τους και τους ε, στερούν βασικά δικαιώματα. Το βλέπουμε στη Βραζίλια με την κυβέρνηση Μπολσονάρου. Έχει περιβαλλοντικά κριτήρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για να επιστρέψει και τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Θα μπορούσα και εγώ να μιλήσω βέβαια και για τις ε, πυρκαγιές στην Εστρεμαδούρα, όπως ε, ε, δεν είναι σίγουρα η μόνη περίπτωση οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Πασκάλ Ντιουράν, επόμενος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω ξεκινώντας από τη σοφόρο τιμή στον Τσίκο Μέντες που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία πριν από 30 χρόνια, που τότε ήδη περασπιζόταν τα δάση του Αμαζονίου και έκτοτε εκατοντάδες ε, συνδικαλιστές και, και ε, αυτόχθονες. Ε, τέσσερις ή πέντε τους τελευταίους μήνες μόλις στη Βραζιλία. Βολσονάρου, Βραζιλιάνικη κυβέρνηση είναι η τέλειοι ένοχοι, ναι, και σίγουρα έχουν ευθύνε. Όμω θέλω να επιμείνω και σε κάτι άλλο η αποψήλωση, αυτά τα εγκλήματα σε βάρος του πλανήτη, της βιοπικιλότητας ε, και των έμβιων όντων, η ερπαγή των γεών ε, και η γενοκτονία δεν έχουν και αυτά ε, αίτιους εδώ στην Ευρώπη. Γιατί να εισάγουμε σόγια για να θρέψουμε το ζωικό μας κεφάλαιο, τα ζώα γιατί ε, εισάγουμε έλαιο. για να πετάνε τα αεροπλάνα μας. Γι' αυτά τους λόγους καταστρέφεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το δευτερόλεπτο στη Βραζιλία. Η μισή αποψήλωση σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται εκεί. Ήρθε η ώρα να δούμε τις δικές μας ευθύνες και όχι απλά να είμαστε θεατές, παθητικοί, ίσως και συνένοχοι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αυτουργοί, συναυτουργοί αυτής της κατάστασης, αυτού του εγκλήματος. Το είπατε, Επίτροπε, σας υποστηρίζουμε. Πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι. Πρέπει να υπάρχει αυτό το καθήκον επαγρύπνησης που θα διέπει τις διεθνείς μας συμφωνίες οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Ναι, εντάξει, να παραμείνουν γιατί θέλουμε να είναι ανοιχτή η Ευρώπη, αλλά διαφορετικά να ε, συντάσσονται αυτέ οι συμφωνίε, να βοηθήσουμε να μην καταστρέφεται ο πλανήτη. Και η συμφωνία Μερκοσούρ δεν είναι κατάλληλη. Πρόεδρο, στείλει μέτσα από του πρασίνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σοκαρισμένη παρακολουθώ την αποδάσωση στον Αμαζόνιο. Το 2020 θα είναι το πιο καταστροφικό έτος στην ιστορία για τον Αμαζόνιο. Η σύμπτωση δε ε, με τον κορονοϊό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον το θέμα, δεν ήταν στο επίκεντρο και σοκαρίστηκα ότι ο Ρικάρντο Σάλλας ήθελε να εκμεταλλευτεί το ότι ο κόσμος ήταν απασχολημένος με την πανδημία για να απλοποιήσει την νομοθεσία. Οι αυτόχθονες πλήττονται σκληρότερα, όχι μόνο γιατί χάνουν τη γη τους λόγω λάθροϊλοτομίας και αρπαγής γης, αλλά και λόγω πανδημίας. Ε, ε, πεθαίνουν δύο φορές περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε έχουν ευθύνη να ε, μην χρηματοδοτούν τους μεγάλους γεωκτήμονες που εκμεταλλεύονται τη γη. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να σταματήσουμε τη συμφωνία με τον Μερκοσούρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χέλμουτ Σόλτς από την ομάδα Γκουε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση Μπολσονάρου κάνει την, έκανε την πρόταση την εξή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα που τα ΜΜΕ ασχολούνται με τον COVID πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να αλλάξουμε τον νόμο. Κλείνει Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό το πνεύμα της κυβέρνησης Μπολσονάρου είναι γεγονός και πράγματι έχετε Κύριε Ντουράντ, έχουμε ευθύνη εάν συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις και συνάψουμε συμφωνία με την κυβέρνηση αυτή η οποία δεν έχει τηρήσει ούτε λέξη από το κεφάλαιο περί βιοπικιλότητας στις υφιστάμενες συμφωνίες. Πρέπει να έχουμε μέσα στην ε, εμπορική μας ε, πολιτική που θα εμποδίζουν ε, αυτά τα εγκλήματα και να είναι επιτέλους δεσμευτικά. Εξάλλου, μπορείτε να υπενθυμίσετε τα όσα έχει υπογράψει ήδη ο κύριος Μπολσονάρο, αλλά αυτός γελάει μαζί μας. χρειαζόμαστε λοιπόν έναν νόμο εδώ πέρα περί εφοδιαστικής αλυσίδας για να απονομώσουμε τα μαύρα πρόβατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Μαρία Αρένα, από Σοσιαλιστές και Δημοκρατίας. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι όσον αφορά την κατάσταση στη Βραζιλία και το θέμα τη αποψίωση των δασών. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με εκείνου που απέκριναν την κυβέρνηση Μπολσονάρου όσον αφορά το μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το μη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το μη σεβασμό τη ε, επικράτειά όσον αφορά την αποψίωση δασών. Αλλά και αυτό που είπε ο Πασκάλ Τιράν με βρίσκει σύμφωνη. Δηλαδή είμαστε και εμεί συνυπεύθυνοι σαν Ευρωπαίοι. Συνυπεύθυνοι που μα οδηγούσε στον τοίχο με εμπορικέ συμφωνίε που απέδειξαν ότι δεν μπορούν είναι ανίκανες να κάνουν σαβαστές τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Κύριε Επίτροπε, όταν λέτε λοιπόν το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη που είναι υποχρεωτική πτυχή σε εμπορικέ συμφωνίε και με το Μερκοσούρ, αλλά όχι μόνο με το Μερκοσούρ, σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε, όταν λέτε ότι αυτά Τυχή θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει. Όχι, αυτό το κεφάλαιο της βιώσιμη ανάπτυξη δεν θεσπίζει, δεν ρυθμίζει τίποτα. Οργανώνει συζητήσει, αλλά δεν επιβάλλει κυρώσει σε περίπτωση μη σεβασμού του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτό που σας ζητάμε δεν είναι marketing. Δεν είναι νέα διατύπωση, νέα γλώσσα, αλλά περιορισμοί, κυρώσεις Λοιπόν, εμπορικέ συμφωνίε. Ναι, αλλά εμπορικέ συμφωνίε που είναι νέα γενιά, αλλά πραγματικά νέα γενιά, που επιτρέπουν πραγματικά να επιβληθούν κυρώσει σε χώρε όπω είναι η Βραζιλία, όπω είναι και άλλε χώρε που δεν τα ε, δικαιώματα αυτά και αυτό το νόμο. Και να υπάρχει και εποπτεία και των πολυεθνικών των Ευρωπαϊκών που όταν επενδύουν σε χώρε που δεν σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν σέβονται τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, να υπάρχει δυνατότητα εκεί τα θύματα να μπορούν να προσφύγουν όπου γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμό αυτού του δικαιώματο καταγγελία. Είναι δικαίωμα ανθρωπότητα. Έχουμε αυτόχθονε πληθυσμού που εξολοθρεύεται στον Αμαζόνιο. Πρέπει να έχει το δικαίωμα πληθυσμό αυτό να μπορεί να καταφύγει, να προσφύγει κατά των πολυεθνικών που δεν σέβονται τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Charles Γκέρεντς από την ομάδα Ρινιό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αποψήλωση των δασών του Αμαζονίου είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που είναι τόσο έρημη όπως είναι αποδασωμένες, αποψηλωμένες αυτές εκτάσεις. Απάζονται γες από ιδιώτες, και που ε, δεν εφαρμόζεται πολιτική, διότι αυτοί που οδηγούν στην επιδείνωση των τασών ξέρουν πολύ καλά ότι μπορούν να βασιστούν στη συνενοχή της κυβερνήσεως και του Προέδρου, του παρόντος. Η πολιτική δεν σέβεται την πολιτική που είχε εφαρμοστεί από το 2004 μέχρι το 2013-2014. Τότε θελοντικά βήματα μείωναν τη ζημιά μέσω ενισχύσεως της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος της Βραζιλίας και μέσω της δημιουργίας ενός ταμείου που είχε σχέδιο, ήταν, ε, ενεταστόταν σαν σχέδιο ετήρησης των δασών. Και η Βραζιλία έχει αναλάβει στην Κοπενχάγη για το κλίμα κάποιες δεσμεύσεις. Πώς να διορθώσουμε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε κάποιες λύσεις, αλλά θεωρώ ότι αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει εθελοντικά να ελέγχουν τις εισαγωγές επιχειρήσεις δεν αρκεί. Και η πολιτική του διαλόγου, ο πολιτικός διάλογος, ναι, πρέπει να γίνεται για να υπάρχει επίγνωση. Αλλά θα προχωρήσουμε πολύ. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει θέση ο Μπολσονάρο. Να θυμηθούμε ότι ανήκει σε αυτού του άνδρες που σε διεθνέ επίπεδο την χάνουν μεγάλη υποστήριξη και με τη βίβλο στο χέρι ε, προσπαθούν να εξαλείψουν ένα, ένα, ένα, ένα τα κεκτημένα τα πολυμερή. Κεκτημένα σημαντικά για την προστασία ε, του, και της ύπαρξης του πλανήτη. Ξέρετε που το πάω στην εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεω Μερκοσούρ, που αν μείνει αμετάβλητη αυτή η συμφωνία, θα την υποδεχτεί ο Μπολσονάρου σαν ένα βραβείο για την ανευθυνότητα. Έτσι θα τη δει. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, Κάρολάιν Ρόουζ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που συμβαίνει στον Αμαζόνιο δεν μπορεί να μας αφήνει αδιαφόρους. Το δάσος του Αμαζονίου είναι κάτι απαραίτητο για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και για την ανθρωπότητα. Διατηρεί, διαφυλάσσει τη βιοπικιλότητα και βιομηχανική καλλιέργεια το καταστρέφει, κυρίως η εντατική καλλιέργεια της σόγιας. Αυτή είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την αποψήλωση των δασών, αλλά και για τη ρήπανση των διαφόρων ποταμών από τα και καταστρέφονται διάφορα ζωικά είδη και αρπάζονται υγιές από τους ε, αγρότες. Διαλύει την προστασία του περιβάλλοντο ο Μπολσονάρου, εκμεταλλεύεται παράνομα ε, τα δάση και αγνοεί τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Δεν είναι μόνο βραζιλιάνικο το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με το Μουρκοσούρ και θέλουμε τη Σόγια, και λέμε στι επιχειρήσει μα που χρηματοδοτούν την καταστροφή, είμαστε συνένοχοι όσον αφορά τη δολοφονία του οικοσυστήματο. Η αλλαγή του κλίματο και η παρούσα κρίση δείχνει ότι τώρα πρέπει να δράσουμε. Η υποψήλωση των δασών συνεχίζει να επιδεινώνεται παρά τον πολλαπλασιασμό των πρωτοβουλειών σε διεθνέ επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί και θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα ισχυρά μέτρα. Αύριο θα είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο Μικ Wallace για την ΚΟΕ. Από το 1970 πάνω 700.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Αμαζονίου έχουν καταστραφεί. Η λεμαργία του αγροτικού τομέα, των μεγάλων επιχειρήσεων και των ε, επιχειρήσεων εξορίξεων και από τι δύο πλευρά του Ατλαντικού οδηγούν στην καταστροφή. Η αλλαγή του κλίματο δεν είναι απειλή για του γεωργού. Οι νεοφιλελεύθερε συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ενώση είναι απειλίε. Έχουμε τη συμφωνία του Μερκοσούρ που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστατεύει συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων να βρούνε τα πιο φθηνέ πρώτε ύλε, αγνώντα το περιβάλλον, το κλίμα ή του αυτόχθονε πληθυσμού. Η συμφωνία του Μερκοσούρ θα οδηγήσει σε περισσότερη υποψήλωση των δασών του Αμαζονίου, θα είναι κάτι κακό για του μικρού καλλιεργητέ στην Ιρλανδία και σε όλη την Ευρώπη όπου ε, δημιουργούμε νέα κυβέρνηση στην Ιρλανδία και το Μερκοσούρ δεν αναφέρθηκε καν στο πρόγραμμα τη νέα κυβέρνηση, που θα γίνει αξιολόγηση, δηλαδή τελικά θα κάνουν τίποτα. Παρά το γεγονό ότι η Φίνα Φόλ και η Πράσινη ήταν αντίθετη πριν από τώρα. Οι μικροί γεωργοί στην Ιρλανδία δεν ανησυχούν μόνο για τη ζωή του, για τη βίωσή του, αλλά έχουν ευαρεθεί από την υποκρισία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και που ζητά τα κάτι μέλη να μειώσουν τι εκπομπέ από τη Γεωργία, προετοιμάζοντα όμω Άγιοι περισσότερα μολυσμένα και περιβαλλοντικά καταστροφικά τρόφιμα και ζωοτροφέ από τη Νότια Αμερική. Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο Μπέρτ Λάγκερ είναι επόμενο από την ομάδα Σοσιαλιστών. Εδώ και δεκαετίες ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό η εμπορική ε, συμφωνία δεν είναι το πιο αποφασιστικό σημείο. Το γεγονό είναι τι πολιτική γίνεται εκεί. Αυτή είναι η ασφαλμένη πολιτική και η πολιτική ε, Μπολσονάρου ε, δυναμτίζει την κατάσταση. Το θέμα είναι πώ θα επιτεθούμε σε αυτό το πρόβλημα, πώ θα μειώσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει και σχέση με το ότι εμείς εισάγουμε πρώτες ύλε από τη Βραζιλία. Κρέας, για παράδειγμα. Και η ζήτηση ε, είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν και να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα της ζήτησης. Και η Επιτροπή ε, δύο χρόνια ε, χρειάστηκε να έχει αυτή την ανακοίνωση προς την αγορά που λέει ότι χρειάζεται πρόσθετα μέτρα ρύθμιση τη ζήτησης ώστε να έχουμε την ε, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού κτλ. Ναι, αλλά τι έγινε μέχρι ε, τώρα, τίποτα. Και θέλουμε δίκαιη, δίκαιη ε, ζήτηση και έγινε μία πρόταση στην έκθεση της συναδέλφου μας για μία λυσίδα εφοδιασμού που θα αξιολογεί ουσιαστικά ε, τα προϊόντα τα οποία θα εισάγουν. Τώρα περιμένουμε τις προτάσεις τις συγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσουμε του χρόνου να έχουμε την νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι μόνο ο Μπολσονάρου. Το 88% των Βραζιλιάνων είναι κατά της ε, ε, αποψήλωσης των δασών όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις. επομένω. πρέπει να τους υποστηρίξουμε και πρέπει να στηρίξουμε και τις περιφερειακές κυβερνήσεις γιατί είναι τελείως διαφορετική θέση τους σε σχέση με αυτή του ε, Μπολσονάρου. Επομένως και η στήριξη των Βραζιλιάνων είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρο, επόμενο ομιλητή Στεφάν Μπιζού από την ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ένα μήνυμα για όλους μας, για τον καθένα μας και την καθεμία μας. Συλλογικά σας ερωτώ. Τι κάνουμε εδώ πέρα εμείς για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ε, πιο δίκαιο, πιο αλληλέγγυο για αύριο που θα βάζει στο επίκεντρο των δράσεών μας ε, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, γιατί μιλάμε για την επιβίωσή μας. Τι νόημα έχουν όλα, στις πόρτες ε, της Ευρώπης της Γαλλικής ε, που είναι ευρωπαϊκό έδαφος δίπλα μας ουσιαστικά στη Βραζιλία έχουμε μια κυβέρνηση της άκρας δεξιάς ε, που εκτελεί ε, με απόλυτη ψυχραιμία και ομότητα ε, ένα σχέδιο καταστροφής ε, του περιβάλλοντος της βιοπικιλότητας, ουσιαστικά κλιματικό σχέδιο και κατά της ανθρωπότητας και των μελλοντικών γενιών. Το έχουμε πει χίλιες φορές και χίλιες φορές έχουμε πέσει στον τοίχο του αλαζονικής, της αλαζονικής υπεροψίας του Μπολσονάρου όλοι μας ε, έχουμε απομονωθεί για ε, να αποφύγουμε την COVID και 115.000 ε, τετραγωνικά μέτρα καταστρέφονταν ταυτόχρονα στην Βραζιλία. Δεν πρέπει να είμαστε συνένοχοι ε, σε αυτό που κάνει η Βραζιλία κατά του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Ε, για να μπορέσουμε να ζήσουμε στο μέλλον πρέπει να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και για να αναπνεύσουμε χρειαζόμαστε δύο πνεύμονες, τον μπλε ε, των θαλασσών, των ωκεανών και τον πράσινο των δασών. Είναι οι μοίρες μας κοινέ το πεπρωμένο μας είναι κοινό όπου και αν ζούμε και γι' αυτό ήρθε η στιγμή να παρέμβουμε. Πριν από πέντε χρόνια μας έλεγαν οι επιστήμονες για το φαινόμενο της πεταλούδας. Ε, αν δεν κάνουμε τίποτα δεν θα υπάρχουν ούτε καν πεταλούδες και ούτε και άνθρωποι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί ο Μάρτιν Χόισλινγκ από τους Πράσινους. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, για κάποια πράγματα δεν θα βρεθεί ποτέ εμβόλιο, όπως η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό πρέπει να ξανάρθουν στο προσκήνιο. Αλλά, εδώ, στη Βραζιλία έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που εκμεταλλεύεται ανέσχυντα την κρίση για να κόψει περισσότερα δάση. Εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και κάποιοι μου λένε ότι συμπεριφέρονται εδώ πέρα σαν να μην υπάρχει καν καταστροφή του περιβάλλοντος στη Βραζιλία. Αν κάνουμε συμφωνία με αυτήν την κυβέρνηση και όποιος κάνει συμφωνία είναι συνυπεύθυνο για την καταστροφή των δασών αλλά και για παραβιάσεις δικαιωμάτων των αυτοχθόνων. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος αγωγέας σόγιας. Η αγροτική μας πολιτική σημαίνει εκτροφή βοηδών με σόγια από Βραζιλία και Αργεντινή. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Λοιπόν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας να βγάλει το θέμα του Μερκοσούρα από την ημερήσια διάταξη και να ασχοληθεί με το κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Η Ιζαμπέλ Σάντος από τους Σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα νούμερα είναι φρικτά. Είχε χαθεί πέρσι ε, μια έκταση ίση με 12.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Φέτος ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Πάνω από 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα η Βραζιλία έχει το 50% της Αμαζονίας. Τι γίνονται λοιπόν εδώ πέρα με το να μην έχουν τους απαραίτητους πόρους οι αρχές δάσο προστασίας σημαίνει ότι κινδυνεύει ο Αμαζόνιος. Και τι γίνεται, ιδιωτικοποιείται επίσης μια τεράστια έκταση γης κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Έχουμε γενοκτονία ή κοκτονία. Αυτά τα έχουν πει οι ηγέτες εκεί πέρα για την τραγωδία η οποία λαμβάνει χώρα η οποία προκύπτει από τις εγκληματικές ενέργειες της κυβέρνησης Μπολσονάρου και έχουν ανέβει εκθετικά οι ανθρωποκτονίες. Οπότε θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Να προστατεύσουμε τα δάση, τους ανθρώπους που ζουν στα δάση και αυτούς που υπερασπίζονται τα δάση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Πράγματι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Το μας φέλετε από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε περίπου 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το χρόνο του μειώνεται το δάσος ε, του Αμαζονίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο και μόνο απορροφά περίπου 500 γήπεδα ποδοσφαίρου σε βόλιο κρέας που παράγεται σε, από δάση που αποψηλώνονται. Στο Μάτο Γκρόσο και μόνο 95% από τα δέντρα που κόβονται για παραγωγή ε, σόγιας ε, γίνονται παράνομα. Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο νόμο, ενθαρρύνει ο Μπολσονάρο την παράνομη άποψη των δασών, ενθαρρύνει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των αυτοχθόνων πληθυσμών. Εμείς στην Ένωση, εμείς είμαστε συνένοχοι. Είμαστε υπεύθυνοι για χιλιάδες εκτάρια, τετραγωνικά χιλιόμετρα αποδάσωση μέσω τη αγωγή βοηού κρέατος και σόγιας και επενδύουμε δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τη μετώπιση αλλαγή του κλίματο. Και επενδύουμε δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε του Ευρωπαίου γεωργού, κυρίω του κτηνοτρόφου βοηθού κρέατο, κατά το του ανταγωνισμού που λαμβάνει η χώρα στι διεθνεί αγορέ. Πώ μπορούμε να εξηγήσουμε λοιπόν το ότι χρησιμοποιούμε εδώ τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματο, αλλά ενθαρρύνουμε την καταστροφή στο εξωτερικό. Αυτή είναι πολιτική Τζέκιλ και Χάιντ. Σταματήστε το Μερκοσούρ και να θέσετε απαγορεύσεις αγωγών σε βόλιο κρέας και σόγια από τη Βραζιλία εδώ και τώρα. Ευχαριστώ. Επόμενος, η κυρία Άβραμ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Λόγω της κρίσης του COVID και λόγω ρήπανσης, εκπληκτικά φαινόμενα ε, συνέβησαν. Ε, λόγω της κρίσεως του κορονοϊού καθάρισε ο αέρας. Στο, στην ατμοσφαιρικό αέρα είδαμε ότι καθάρισε και στα ποτάμια μας είδαμε διάφορα είδη που δεν είδαμε εδώ ε, και χρόνια. Και έχουμε δει ελάφια να μπαίνουν στις πόλεις. Ε, δείχνει τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το 2050. Είναι μια πρόβα αυτή από τη στιγμή που θα εφαρμόσουμε το σύμφωνο το πράσινο. Επίσης, είδαμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Στον Αμαζόνιο, στην περιοχή του Αμαζονίου, 50% περισσότερα δέντρα κόπηκαν από παραπάνω από ό,τι πέρσι την ίδια περίοδο. Και η τάση της παράνομης υλοτομίας ε, συνεχίζεται να αυξάνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την αισιοδοξία μας όσον αφορά τη σωστή συμπεριφορά κάποιων κρατών που θέλουμε να έχουμε ως εταίρους και θα πρέπει να επιβάλλουμε πιο αυστηρούς όρους στις διαπραγματεύσεις μας και στις εισαγωγές μας. Σαν εισηγήτρια σκιώδης για την νέα για τα δάση, ξέρω ποιες προσπάθειες καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σέβονται όλους τους όρους του οικολογικού συμφώνου. Αν δεν επιβάλλουμε τους ίδιους όρους όμως τους άλλους, όχι μόνο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την αποψήλωση των δασών στον Αμαζόνιο, αλλά θα επιβάλλουμε αθέμητο ανταγωνισμό και θα χάσουμε. Το πράσινο σύμφωνο ε, είναι δικό μας, δεν πρέπει να αφορά μόνο εμάς. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Πρασίνων, ο κύριος Χόγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Λέει ο κόσμος ότι ο Αμαζόνιος είναι ο πνεύμονας, είναι οι πνεύμονες του πλανήτη. Αλλά το αντίθετο των πνευμόνων είναι απορροφά περις πολύ διοξίδιο του άνθρακος. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι του πλανητικού συστήματος. Εγώ είμαι μετεωρολόγος και πρέπει να πω ότι ξέρουμε τι απειλή θα είναι για μας εάν συνεχίσουμε να χάνουμε ε, το δάσος ε, του Αμαζονίου. Είναι πολύ σημαντικά τα δάση του Αμαζονίου για το παγκόσμιο κλίμα. Αυτό δεν είναι κάτι συζητήσιμο. Είναι γεγονός, επιστημονικό γεγονός. Οποιοςδήποτε στην αίθουσα εδώ πιστεύει ότι οι οικονομικές πτυχές θα πρέπει να υπερτερούν των άλλων, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι θα μπορείτε να αναπνεύσετε με, και να εισπνέετε ετήσια λογιστικά, ετήσια εκθέσει. εκθέσεις. Νομίζω ότι θα μπορείτε να θραφείτε με χρήμα. Αν όχι, βοηθήστε να πολεμήσουμε όλοι ούτως ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Επίτροπος, ο κ. έχει το λόγο, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ευρωβουλευτέ. νομίζω ότι είναι σαφέ το μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα. Η αντιμετώπιση της αποψήλωση του δάσου του Αμαζονίου είναι προτεραιότητα μεταξύ σχεδόν όλων ε, στο πολιτικό φάσμα. Και νομίζω ότι έδειξε πως ε, είναι σαφές και κατανοητό ότι πρόκειται για πολυσχηδείς προκλήσεις για την ε, περιοχή του Αμαζονίου. Φυσική, πόρη και πληθυσμός. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά με ολιστικό τρόπο στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής. Κυρία Μακίνες, πολύ σωστά είπε ότι πρέπει να δούμε πόσο πολύπλοκη είναι η λυσίδα φωδιασμού. Αυτό είναι αληθε. και είναι κάτι ε, που συνιστά πρόκληση για εμά. Αυτό κάνουμε όμω. Σα διαβεβαιώ. Συνεργάζομαι στενά με όλου του συναδέλφους ώστε τις περιβαλλοντικές, τις γεωργικές, τις εμπορικές, υγειονομικές, κλιματικές πτυχές να τις ε, εξετάσουμε από κοινού και σε συνδυασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα διαβεβαιώ ότι δεν δίνει μόνο σημαντική τεχνική και οικονομική υποστήριξη στι χώρε για να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει αυτέ, αλλά και ακούμε πολύ προσεκτικά τους αυτόχθονες που πλήττονται άμεσα. Και όπως και η κυρία Μπούρκχαρτ και η κυρία Ματίας. Και τις ε, ε, χώρες πολιτικές εξετάζουμε για να μειωθεί της Ένωσης το αποτύπωμα σε στενή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα και διάβλους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Επίσης, αναλαμβάνουμε δράση για να στηρίξουμε παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της αποδάσωσης και για την προστασία των δικαιωμάτων των τοπικών κοινωνιών ε, και των αυτοκτόνων που κινδυνεύουν λόγω της αρπαγής γης και της αποψήλωσης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσβλέπω και στο αποτέλεσμα των ε, συζητήσεων που θα έχετε επί της εκθέσεως νομοθετικού περιεχομένου της κυρίας Μπούρκχαρτ για το πώς μπορούμε να ε, αναστρέψουμε το φαινόμενο της ε, αποψήλωσης. Έχουμε την COP26 στην Γλασκόβη και στο Κομίνγκ και αυτές οι κομβικές ε, συναντήσεις κορυφής θα είναι πάρα πολύ αποφασιστική σημασία. Πρέπει να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε κρίσιμα οικοσυστήματα όπως είναι τα δάση. Δεν είναι αυτό μόνο μια λύση για την πρόσταση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Πολύ μιλήσατε για την ε, κυβέρνηση της Βραζιλίας εμείς. Καλούμε τις εθνικές αρχές και τις βραζιλιάνικες επομένω να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να αντιμετωπίσουν την αποψήλωση των δασών για διεθνή και περιφερειακή συνεργασία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τεχνική υποστήριξη ώστε να μειωθεί γρήγορα η αποψήλωση αλλά και με βιώσιμο τρόπο. Θέλουμε όμως να δούμε και σαφή προθυμία και από την άλλη πλευρά. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Στεφανούτα, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι το πρόβλημα της αποψήλωσης των δασών δεν υπάρχει μόνο στο εξωτερικό, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από πολύ κοντά παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Ευρώπη και είμαι αποφασισμένος να πάρω και εδώ πολύ αυστηρά δραστικά μέτρα. Επειδή επίση πολύ αναφερθήκατε στι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου, θέλω να επενθυμίσω πως όλες οι σύγχρονες εμπορικέ μα συμφωνίες περιλαμβάνουν φιλόδοξες ρήτρε. Μπορεί να είναι ε, ακόμα ε, ατελείς και να επιδέχονται βελτίωση, αλλά μιλούμε για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και εφορία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνίε με τι χώρε Μερκοσούρ, ε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε όλε τι πολιτικέ των χωρών σε όλου του τομεί επειδή συνάπτουμε αυτή τη συμφωνία. Φυσικά και όχι. Όμω ε, είναι ένα τρόπο αυτό να ε, έχουμε αμοιβαιότητα και ανάληψη δεσμεύσεων. Είναι ένας τρόπος να έχουμε διάλογο και συνεργασία με τη Βραζιλία και τις άλλες χώρες περιοχές για να τις πιέσουμε και να τις ενθαρρύνουμε, τις παροτρύνουμε να τηρήσουν τι δεσμεύσει που ανέλαβαν από κοινού μαζί μα στη Συμφωνία των Παρισιών. Επίση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα επεξεργαζόμαστε. Χώρε η Μερκοσούρ, που μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, περιλαμβάνουν δεσμεύσει κατά τη αποψήλωση στι υποσχέσει που έδωσαν στο πλαίσιο και στι δεσμεύσει που έδωσαν στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρισίων. Και για τη συσκευασία των ε, κρεάτων Υπάρχει αυτό το μαρτώριο για τη Σόγια και οι ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Θα παρακολουθούμε όλα αυτά και για να ολοκληρώσω, ναι, σίγουρα παραμένει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και σίγουρα θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε την νομοθετική αυτή πρόταση που θα σας καταθέσουμε του χρόνου. Θα συνεργαστώ στο μέλλον μαζί σας όπως μέχρι τώρα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ, η Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση εδώ Ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας στην 1 και 30 το μεσημέρι.